Καλημέρα σας. Άρχεται η πρωινή συνεδρίαση. Η μέσα διάταξη προβλέπει την κοινή συζήτηση σχετικά με τα δραστηριότητες πιστοτικών ενδυμάτων και νευροπτική. Ε, προληπτική συγγνώμη εποπτεία, πιστοτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων ε, του κυρίου Κάρα. Δίνω τον ε, λόγο στον κύριο Κάρα Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε,